Βάσει το 216, σημείο 4 του κανισμού θα ήθελα να σας πω ότι οι διορθώσεις που κατατέθηκαν ε, χθες ε, μέχρι τις 5 η ώρα ε, εγκρίνονται, εφόσον δεν αμφισβητήθηκαν, θεωρούνται οι διορθώσεις αυτές αποδεκτές. Από την ΚΟΕ έχω πάρει μία πρόταση να...